την προσάρτησε ε, στα συμπεράσματα σχετικά με τα αποτελέσματα όσον αφορά στους στόχους της χιλιετίας για την ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτροπε. Ευχαριστώ την κυρία Θεοχάρους. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ και τους διερμηνείς. Λύεται η συνεδρίαση αύριο το πρωί, συνεχίζει η Ολομέλεια στις 9 το πρωί. Ευχαριστώ πολύ.